Oh, I'm, I Πούμε πάρα πολύ ότι χάσαμε κάποιους συναδέλφους που απουσιάζουν, πήγανε για καφεδάκι ή για κάποια ιδιωτική υπόθεση. Κάποιοι είναι παρόντες και γι' αυτό πιστεύω θα έπρεπε να ξεκινήσουμε ευχόμενοι ένα, μια καλή, ένα καλό απόγευμα συνεδρίασης. Θα επανέλθουμε. Έχουμε την έγκριση της, του σχεδίου ημερήσιας διάταξης. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνεται λοιπόν και για ανακοινώσεις Προέδρου δεν έχω διάφορα, κανείς δεν έχει ζητήσει κάτι και τώρα είμαστε στο σημείο 5 παρουσίαση της ε, Ombudsman <clears throat> της ε, ετήσιας ε, έκθεσης από πλευρά τη. Έμιλη, είναι ιδιαίτερη χαρά, Έμιλη Ωρέλη, που να σας έχουμε στην κοινοβουλευτική μας επιτροπή από κοινού εδώ σε εμά. Έχετε τον λόγο λοιπόν να μας προσφωνήσετε Εμίλιο Ρέλη. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Βίξτρομ. Καλό σας απόγευμα σε όλους σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω την ετήσια έκθεση για το 2015 σε εσά. Να παρουσιάσω το έργο που, με το οποίο ασχολούμαι από την επανεκλογή μου ως ε, συνηγόρου διαμεσολαβητού από το 2014. Εργαζόμαστε σε πολλά μέτωπα εσωτερικά προσπαθώντας σε σχέση με τα θέματα αυτά να είμαστε ακόμα πιο αποτελεσματικοί ώστε τα παράπονα και τα κύματα των πολιτών να μπορούν άμεσα να διευθετούν, να διεκπεραιώνονται και στις ε, ε, έρευνες που κάνουμε για να μπορέσουμε να συλλέξουμε στοιχεία και πιο σημαντικό να συνεργαζόμαστε με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ε, Διαμεσολαβητών ή Συνηγόρων που έχω την τιμή να προεδρεύω αυτού να έχουμε πρόσθετη αξία και στο δικό μας έργο και του θεσμικού οργάνου και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητού και όσον αφορά τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες. Γενικά αυτά με την πρώτη διαφάνεια κιόλα, 250 εξετάσεις γίνονται τήσια μάλιστα με ε, συστημική και στρατηγική ε, μορφή στο χαρακτήρα που εντάσσουμε μέσα σε μια εξεταστική δράση αρκετά θέματα παραφώνων. Ο μεγαλύτερος πελάτης μας είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εδώ σε σχέση με την, τις ιδιαίτερα υψηλές προδιαγραφές που διέπουν την διοίκηση και διαχείριση από πλευρά της είναι όμως το πιο σημαντικό θεσμικό όργανο για τους πολίτες. Έχουμε και άλλα θεσμικά όργανα όπως το Ευρωκοινοβούλιο όσον αφορά το διοικητικό έργο, την ΕΦΣΑ που είναι ένα σημαντικό θεσμικό όργανο για μας επειδή εκατοντάδες, χιλιάδες άτομα υποβάλλουν αίτηση για να απασχοληθούν στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και αν θεωρηθεί ότι δεν έτυχαν θεμητής σωστής αντιμετώπισης μπορούν να προσφύγουν σε εμά και να υποβάλουν παράπονα θέματα τα οποία εξετάζονται και όσον αφορά ισχυρισμού ε, διαφθοράς για παράδειγμα περιπτώσεων διαφθοράς ε, όπου εξετάζονται το τι έχει πράξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλοι για να ε, αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό και αν ή είμαστε ικανοποιημένοι με τις απαντήσεις. Όλα αυτά συσχετίζονται και με τα θέματα που η Όλαφ επιλαμβάνεται αυτών και σε σχέση με όσους ε, εμπλέκονται σε σχέση με τις εξεταστικές δράσεις, ώστε να είναι πλήρως νόμιμες και ευθυγραμμίζονται με τα όσα πρέπει να γίνονται. Η επόμενη διαφάνεια αφορά τα κυριότερα σημεία, τους κυριότερους τομείς ε, όσον αφορά τους τελευταίους μήνες. Για παράδειγμα, Ιανουάριο τις εκθέσεις ομάδων πραγματογνωμόνων που ολοκληρώνονται και κατέβαλε προσπάθεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη τις συστάσεις και να υπάρξει επιτήρηση πόσο όλα αυτά υλοποιούνται κατά τους επόμενους μήνες και όσον αφορά την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ώστε συλλογικά να μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο το Φεβρουάριο και εδώ σε σχέση με την δική μας έρευνα όσον αφορά τους πληροφοριοδότες και είχαμε το θέμα ότι δύο μόνο θεσμικά όργανα είχαν υιοθετήσει διατάξεις για τους πληροφοριοδότες και τώρα μπορούμε να πούμε ότι όλα τα θεσμικά όργανα έχουν υιοθετήσει διατάξεις για τους πληροφοριοδότες. Αυτό είναι πολύ θετικό διότι και πάλι όπως έχετε συνειδητοποιήσει αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Έχουμε μια υποεξέλιξη ομάδα εργασίας ε, το Μάρτιο για την TTIP και τη διαφάνεια των διαδικασιών της διατλαντικής αυτής συμφωνίας εμπορίου και επενδύσεων. Κοινοβουλευτική Επιτροπή πάμπολοι εμπλέκονται στο θέμα των διαπραγματεύσεων και όσο ήταν δυνατόν να γίνει αυτό. Είναι λοιπόν πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα οι εμπορικές διαπραγματεύσεις ε, που πρέπει να ε, καλύπτονται. Ικανοποιήθηκα με την πρόοδο που επετεύχθη από την Επιτροπή όσον αφορά την διαφάνεια σε σχέση με την TTIP τον Απρίλιο. Είχαμε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο του Σεμιναρίου Ombudsman στη Βασοβία στέφθηκε με επιτυχία αυτό το εγχείρημα και κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης αντί να γίνεται σε ένα κράτος μέλος και να εξετάζουμε το συγκεκριμένο ρόλο του Ευρωπαίου διαμεσολαβητή ε, φέτος θα γίνει στις Βρυξέλλες πράγμα το οποίο μόλις ε, αποφασίστηκε η ιδέα είναι τα κράτη-μέλη και από πλευράς ομπούτσμεν να ευαισθητοποιηθούν πολύ περισσότερο για το θεσμικό έργο στο οποίο εμπλέκονται τα θεσμικά όργανα και το Κοινοβούλιο τον Μάιο εκδήλωση για την ε, διαφάνεια όσον αφορά το λόμπινγκ για τη διαφάνεια και με συμμετοχή του Επιτρόπου Τίμερμανς ε, ιδιαίτερα όσον αφορά τις πληρωμές για μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και τις δράσεις της Επιτροπής υπέρ αυτών τον Ιούλιο πολύ σύντομα τώρα έχουμε την Ad hoc Ηθική Επιτροπή όσον αφορά τις συστάσεις ε, ώστε ενεργώς να δημοσιοποιούνται οι διαδικασίες σε σχέση με τη λογοδότηση ή την αναφορά σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν ε, από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τις δραστηριότητες ε, των ταχυδρομείων. Εξετάζονται αυτά τα θέματα από την Επιτροπή έχουμε τον Αύγουστο την ε, επανεξέταση της εφαρμογής ε, της σύμβασης και των διατάξεων των δικαιωμάτων των ατόμων με ειδικέ ανάγκες και αυτό είναι υποεξέλιξη έργο. Δεν εμπλέκεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο περαιτέρω και αυτό αφήνει τον διαμεσολαβητή και την, ε, το Σύλλογο για τα Δικαιώματα των Ατόμων με ειδικέ Ανάγκες, με μειονεξίες. Εξετάζουμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα ώστε με τον καλύτερο τρόπο να υλοποιείται αυτή η σύμβαση που έχει πάρα πολύ σημαντικό χαρακτήρα για αυτά τα άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Σεπτέμβριο μια άλλη εκδήλωση για τον τριμερή διάλογο ή τρίλογο που θα ολοκληρωθεί και θα υποβληθούν και προτάσεις προς τα θεσμικά όργανα για το πώς αυτό το συγκεκριμένο θέμα, πώς οι τριμερείς διάλογοι μπορούν να καταστούν πιο διαφανείς για τους πολίτες και να, ενθυμούμαστε, να ότι πρέπει να υπάρξει ευαισθητοποίηση όσον αφορά τους πολίτες για αυτά τα θέματα τον Οκτώβριο, συστάσεις όσον αφορά τη διαφάνεια για το, τους λομπιίστες ε, των καπνοβιομηχανιών και εμπόρων καπνού είναι κάτι που ελπίζω ότι έγκαιρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να επανέλθει σε αυτό σε σχέση με τις συστάσεις ώστε ενεργά να μπορέσουν να δημοσιοποιηθούν τα όσα τεκταίνονται σε σχέση με τις καπνοβιομηχανίες στα κράτη-μέλη, ώστε να ευθυγραμμιζόμαστε σε σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών ε, για την αντιμετώπιση του καπνού και του καπνίσματος. Και είναι πάλι κάτι το οποίο πρέπει να θυμόμαστε. τον Νοέμβριο Ήμουν πάρα πολύ υπερήφανη για το ότι μπορέσαμε να ε, αναλάβουμε αυτή τη δραστηριότητα και από πλευράς ε, Προεδρίας. Ε, ήταν μια πολύ επιτυχή συγκυρία και μπορούμε έτσι να στραφούμε και στην επόμενη δεκαετία και περαιτέρω αυτής το Δεκέμβριο μια άλλη σημαντική επιτυχία για την υπηρεσία μας. Αρχίσαμε τις εργασίες ε, για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τους κανόνες και κανονισμούς για τη διαφάνεια και την εμπλοκή της με τους ε, ε, ενδιαφερόμενους και όσους συμμετέχουν. Ιδιαίτερα όσον αφορά τα αποτελέσματα των ανακοινώσεων από πλευράς ε, Προέδρου της Κεντρικής, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τους κανόνες και κανονισμούς, ώστε κανείς να μην έχει συγκεκριμένα προνόμια προτερήματα όσον αφορά τις συναλλαγές του ε, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναγνωρίζοντας ε, ότι είναι όλο και πιο σημαντικός ο ρόλος της σε σχέση με τις δραστηριότητες αυτές. Ήταν μια πολύ θετική έκβαση. Αυτά είναι παραδείγματα και ε, συνηθισμένων παραπονών που υποβάλλονται όπως το 2015. Ένα, να ε, μπορέσετε να έχετε μια γεύση για το τι συμβαίνει όπως και την Επιστημονική Επιτροπή για τα Γενετικά Τροποποιημένα ο, επίσης σε σχέση με τα κονδύλια που διανέμονται όσον αφορά την έρευνα ε, καθυστερήσεις όσον αφορά την ε, αντιμετώπιση ε, παραπόνων και προσφυγών για παραβιάσεις και παραβάσεις πρόσβαση στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων όσον αφορά θέματα φοροδιαφυγής. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα για τέτοιου είδους παράπονα. Αυτά όσον αφορά τις θεσμικές μας σχέσεις που ήταν ιδιαίτερα θετικές δεν είναι μόνο το ότι εμπλεκόμεθα με ένα θεσμικό όργανο όταν υπάρχει κάποιο παράπονο. Είναι θετικό να έχουμε σε όλα τα επίπεδα σχέσεις θεσμικές και στο επίπεδο γραμματιών και διευθύνσεων ώστε να υπάρχουν άτυπες και επισημοποιημένες σχέσεις και επαφές μαζί τους με τα θεσμικά όργανα. Αυτή είναι μια άλλη επιτυχία από πλευρά μας όπου συμφώνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθηθεί η διαφάνεια της αρχής του revolving door ε, της ε, ανακύκλωσης ας το αποκαλέσουμε έτσι άρχισε σε μια ετήσια βάση να γίνεται αυτό ε, και αυτά σε σχέση με τα στοιχεία για τα άτομα τους προηγούμενους ανώτερους αξιωματούχους ε, που εγκατέλειψαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άρχισαν να εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Και σε τι ε, πρόκειται να εργαστούν ε, οι λεπτομέρειες που σε πολύ περιορισμένο πλαίσιο γνωστοποιούνται. Νομίζω μπορεί να βελτιωθεί αυτό το πλαίσιο και να γίνεται αυτή η πληροφόρηση σε μια πιο τακτική βάση. Και να δούμε και το θέμα των ανώτερων αυτών αξιωματούχων και τα ονόματα του αν θα δημοσιοποιούνται ή όχι, διότι υπάρχει αυτή η σημαντική πτυχή που πρέπει να επιληφθούμε αυτής. Χαίρομαι λοιπόν το ότι έχει προαχθεί και αυτό. Και τώρα για το επόμενο, και αυτό πάλι είναι η πρώτη περίπτωση παράλληλων ε, εξεταστικών ενεργειών και το τι πρέπει να γίνει σε σχέση με την ε, κοινότητα και τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και τα θεσμικά όργανα, αν υπάρχει ένα θέμα το οποίο ε, δημιουργεί ε, κάποια ζητήματα. Αν εμείς ε, συλλογικά μπορέσουμε να εμπλακούμε και συμμετάσχουμε, τότε μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη απήχηση και στα θεσμικά όργανα και σε σχέση με τα κρατη Αυτό αφορά τις κοινέ δράσεις επιστροφών που συντονίζει η Frontex σε σχέση με τον έλεγχο συνόρων όσον αφορά ετούντες άσυλο, και το πόσα, πόσα άτομα μπορούν να επιστραφούν σε τρίτες χώρες, σε άλλες χώρες. Κάποια κράτη-μέλη έχουν προχωρήσει σε σχέση με αυτό αλλά άλλοι διαμεσολαβητές δεν γνώριζαν για τον ρόλο που ε, μπορούσαν να έχουν από ένα σύνολο 19 σε σχέση με τις ε, εκθέσεις ε, που συντάσσονται για το τι συμβαίνει στα κράτη αυτά. Η Frontex πολλές από τις συστάσεις τις έλαβε υπόψη και υπάρχουν και πρακτικά θέματα αντιμετώπιση παιδιών και γυναικών για παράδειγμα και το τι συμβαίνει όταν επιστρέφουν κάποια άτομα και να υπάρχουν ρήτρες ασφάλειας ότι θα αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια με τον δέοντα τρόπο αυτοί οι άνθρωποι διότι υπάρχουν και αλλαγές και διαφορές και θα πρέπει εδώ μέσα στο πλαίσιο αυτών των περιοριστικών όρων, να δούμε τι μπορεί να γίνει και για την Frontex που μπορεί να μην έχει την άμεση ευθύνη όσον αφορά την, τα θέματα αυτά εναντί κρατών μελών και είναι συντονιστικό ε, το έργο τους. Θα πρέπει τουλάχιστον να διασφαλίζεται ότι θα είναι η βέλτιστη μεταχείριση που θα διασφαλίζεται στα άτομα αυτά μέσα από αυτές τις ε, διαδικασίες. Και πάλι επανέρχομαι σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών, μια μεγάλη σύνοδος τον Ιούνιο 2016 στις Βρυξέλλες, όπου πολλοί ήταν, μπόρεσαν να συμμετάσχουν και να προσφωνήσουν. Τρία θέματα, η μεταναστευτική κρίση, <clears throat> η διαφάνεια σε σχέση με λομπιίστες και το κράτος δικαίου και η Frontex όπως και ανώτεροι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρακολούθησαν ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να δείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση το ευδιάκριτα το πρόσωπό της ότι δεν είναι κάποια πρόσωποι γραφειοκράτες αλλά είναι άνθρωποι που επομίζονται αυτό το πάρα πολύ ε, υψηλού επίπεδου έργο ε, που πρέπει να επιτελεστεί από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμμόρφωση τώρα με τις προτάσεις μου όσον αφορά συστάσεις του 2014. Πάνω από το 80% φτάσαμε στο 90% υιοθέτησης και συμμόρφωσης. Έχουμε όμως σε κάποια πεδία μη συμμόρφωση ακόμα. Πρέπει να πούμε ότι γενικά από πλευράς ε, της ε, πείρας μου μπορούσα να δω και, να, ε, και βίωσα ότι από πλευράς υψηλότερης αποδοχής των συστάσεων και σε σχέση με την δραστηριότητά του σε ένα κράτος μέλος ή σε μια περιφέρεια για το θέμα του κράτους δικαίου και των διεργασιών όταν αυτά τα λάμβαναν ιδιαίτερα σοβαρά υπόψη όλοι συμφώνησαν να σεβαστούν τους κανόνες του παιχνιδιού και όλοι αναγνώρισαν τη σπουδαιότητα του ρόλου του διαμεσολαβητή σε σχέση με τα κράτη-μέλη και όλα αυτά δείχνουν ότι γενικά ε, από πλευράς θεσμικών οργάνων. Τα θεσμικά όργανα πράγματι ε, ευθυγραμμίζονται και συμμορφώνονται με τις συστάσεις όσον αφορά τον ρόλο του διαμεσολαβητή και τις ε, διατάξεις ελέγχου που πρέπει να διασφαλίζονται τι θα ακολουθήσει ολοκληρώνοντας το έργο μας σε σχέση με τους ε, τριμερείς διαλόγους ε, για την ε, διαφάνεια, εξετάζοντας τι μπορεί να γίνει με τους ειδικού συμβούλους και σε σχέση και με, την, με ισχυρισμούς για, την, για αντικρουόμενα συμφέροντα, θα δούμε πώς θα διασφαλιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτοί οι κανόνες και κανονισμοί θα είναι σεβαστοί και σε σχέση με το διορισμό τέτοιων συμβούλων όμως είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη το θέμα συμβούλων διότι είναι ε, εξέχουσες προσωπικότητες ε, πραγματογνώμονες ε, σε σχέση με τα θέματά τους και δεν θα πρέπει σε σχέση με θέματα τα οποία από πλευράς ε, Επιτροπής ε, ε, δεν θα έπρεπε να αποτελούν πρόσκομα, να μπορούν να εξετάζουν τη δυνατότητα αυτή να συμμετέχουν. Άτομα δηλαδή που θα συμμετέχουν στην δραστηριότητα αυτή συμβούλων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το έργο. Διαφάνεια λοιπόν και από πλευράς του Συμβουλίου είναι κάτι το οποίο πρέπει να διασφαλιστεί ώστε σε σχέση με τα παράπονα που υπάρχουν να υπάρξει συνειδητοποίηση αυτών των θεμάτων, να είναι γνωστό το τι είναι, ποια είναι τα θέματα που δημιουργούν ε, τριβές και πώς μπορούν να αρχίσουν να διευθετούνται ή να διασφαλίζεται μεγαλύτερη διαφάνεια. Ξεκινήσαμε θετικά νομίζω σε σχέση με την Ευρωομάδα Eurogroup και σε σχέση και με τον κύριο Dijsselbloem που ανέλαβε την Προεδρία και την ε, δημιουργία, προσπάθεια δημιουργίας ε, πλαισίου διαφάνειας όσον αφορά την ε, Ευρωομάδα, το Eurogroup. Τουλάχιστον αυτό είναι η εντύπωση που διαχέεται σε σχέση και με τους πολίτες. Υπάρχει εδώ ιδιαίτερη ευθύνη να διασφαλίζεται η διαφάνεια. Ήταν καλή λοιπόν θετική ανταπόκριση και έχει δεσμευτεί το πλαίσιο αυτό να διασφαλίζει ακόμα μεγαλύτερη διαφάνεια σε σχέση με το έργο που επιτελείται. Πρέπει να δοθεί συνέχεια σε αυτό και για την Κορεπέρ. Επίσης σημαντικό το θέμα και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι μέσω των ε, αντιπροσώπων ε, και η εμπλοκή της Επιτροπής ε, ε, των εκπροσώπων θα μπορεί να διασφαλίσει. Είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη το ότι από πλευρά σας τελεχών και σε σχέση με την, ε, το έργο που επομιζόμαστε να δούμε ποιος είναι ο ρόλος μας, πώς μπορούμε να δράσουμε και τι είναι δυνατόν να γίνει. Χρειαζόμαστε όλοι να μπορούν να συμμετάσχουν και να προχωρήσει αυτό το εγχείρημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για την πολύ πλήρη παρουσίασή σας. Να υπενθυμίσουμε ότι το 2015 είχαμε την 20η επέτειο της δημιουργίας της θέσης του διαμεσολαβητή. Όλα αυτά που ακούσαμε ε, δείχνουν την επιτυχία της θέσης αυτής. Ε, συνεχίζεται τώρα, ενώ, και ενώ διανύουμε το 21ο έτος ε, από τη δημιουργία της θέσης, συνεχίζουμε αυτή την επιτυχημένη δραστηριότητα. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Μαριά, στον εισηγητή της Επιτροπής μας. Ε, Ευχαριστώ. Καλωσορίζω την Ευρωπαία Διεμεσολαβήτρια στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών. Τη συγχαίρω για τη θαυμάσια δουλειά που κάνει. Και επιτρέψτε μου να συνεχίσω την ομιλία μου στα ελληνικά. Είναι ιδιαίτερη χαρά να, που έχω αναλάβει ως ραπορτέρ ε, για την ε, δράση της ε, Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας και θα έλεγα πρώτα απ' όλα έχουμε δύο σημαντικές εκθέσεις προηγουμένως που υπάρχουν. Πρώτα απ' όλα του συναδέλφου Βαλέσα και της ε, κυρίας Καμπεσόν που έκαναν τις αναφορές τους και τις εκθέσεις τους τα προηγούμενα χρόνια. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή δουλειά που έχει γίνει και έχουμε δύο σημαντικά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του θέματος αυτού. Επομένως θα μπορούσαμε να έχουμε αυτά ως μια σημαντική βάση. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε μια ε, δουλειά που έχει γίνει από την πλευρά της Ευρωπαίας ε, Διαμεσολαβήτριας, η οποία έχει θέσει πάρα πολλά σημαντικά ζητήματα, στα οποία μάλιστα αναφέρθηκε εκτεταμένα. Και είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα γιατί 22 χρόνια μετά από την έκδοση του βιβλίου μου The European Ombudsman που είχα την ευκαιρία να εκδώσω στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης έχω την ευκαιρία να Λέω ως Ευρωβουλευτής να εισηγηθώ μια έκθεση εδώ στους ε, συναδέλφους με σημαντικές παρατηρήσεις. Και χαίρομαι διότι ένα από τα θέματα που είχα επεξεργαστεί πριν από 22 χρόνια είναι ο έλεγχος της διακριτικής ευχέρειας της Κομισιόν. Αν η Κομισιόν δηλαδή, ενεργώντας με το άρθρο 169, δηλαδή όταν υπάρχει μια παραβίαση εκ μέρου ενό κράτου μέλου τη νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει και στην παραπομπή τη υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Διότι η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ήταν ξεκάθαρη ότι υπάρχει μια πλήρη διακριτική ευχέρεια σε επίπεδο Κομισιόν. Είχα υποστηρίξει τότε σε ένα άρθρο μου ότι υπό όρου και προποθέσει ενδεχόμενα η μη παραπομπή μια υπόθεση από πλευράς Κομισιόν με βάση το άρθρο 169 στο δικαστήριο ενδεχόμενα να αποτελεί περίπτωση κακοδιοίκηση. Χαίρομαι λοιπόν που βλέπω φέτος ότι υπάρχει μια τέτοια απόφαση από την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια στο θέμα αυτό και έτσι φαίνεται πώς μπορεί κανείς όταν είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο ή ερευνητής να εκφράσει ελεύθερες σκέψεις με προτάσεις οι οποίες έρχονται πολλέ φορέ μετά από πολλά χρόνια το πλήρωμα του χρόνου να γίνουν αποδεκτέ. Θέλω να πω δηλαδή ότι η εργασία που γίνεται από πλευρά τη Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας είναι πάρα πολύ σημαντική. Και α έρθουμε λοιπόν στο πρώτο θέμα που ονομάζεται διαφάνεια. Αυτό το θέμα που είναι καθοριστικό για τη δουλειά που κάνει ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Θεωρώ σημαντική την δραστηριότητα και την πρωτοβουλία που πήρε η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια στην TTIP. Διότι αυτό είναι ένα θέμα που απασχόλησε τους βουλευτές, απασχόλησε την Επιτροπή μας με πάρα πολλές αναφορές, απασχόλησε ε, την κοινωνία των πολιτών. Και νομίζω ότι οι ενέργειες που έκανε η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, και αυτό το είπα την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο που συζητούσαμε τα θέματα διαφάνειας, η δουλειά που έκανε και η πίεση που άσκησε ε, στην Κομισιόν μαζί και με τους Ευρωβουλευτές έφεραν ένα πρώτο αποτέλεσμα να έρχεται πλέον η Κομισιόν και να έχει μια μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαπραγμάτευση για την TTIP. Όμως πρέπει πολλά πράγματα στο θέμα της TTIP να γίνουν και να συνεχιστούν. Το θέμα της διαφάνειας αφορά επίσης και τον τρίλογο, δηλαδή τη συζήτηση που γίνεται για την ε, διαμόρφωση προτάσεων μεταξύ των τριών οργάνων. Και αυτό είναι πολύ σημαντική δουλειά που έχει κάνει επίσης η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια. Υπάρχουν φυσικά και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όργανα που λειτουργούν ad hoc στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εκφεύγουν μέχρι στιγμής του ελέγχου, όπως είναι το Eurogroup. Διότι το Eurogroup αυτή τη στιγμή παίζει τεράστιο σημαντικό ρόλο λαμβάνει αποφάσεις οι οποίες επηρεάζουν την οικονομική λειτουργία όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λαμβάνει αποφάσεις ιδίως με μέτρα σκληρής δημοσιονομικής πολιτικής που επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία της ζωής των πολιτών. Και πολλές από αυτές τις αποφάσεις, κατά την άποψή μου, ε, άπτονται και παραβιάζουν πολλές φορές και τα δικαιώματα των πολιτών. Και είναι ένα θέμα που το συζητήσαμε στην έκθεση για την εφαρμογή ανθρωπίν, του χάρτη ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί υπάρχει μια ολόκληρη παράγραφος ε, στη μελέτη ότι η Τρόικα, δηλαδή το, η ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν παίρνουν μέτρα στο πλαίσιο των προγραμμάτων ε, προσαρμογής των μνημονίων πολλές φορές ε, παραβιάζουν το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτό είναι κάτι σημαντικό που πρέπει να το δούμε και σε σχέση με το Eurogroup. I will be very brief, I will finish in, if I have one minute. Okay. Δώστε μου ακόμα ένα λεπτό. Ενός, το θέμα του ελέγχου του Eurogroup της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να δούμε επίσης αν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων κατά τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως μέλος της Τρόικας και ως ανεξάρτητης νομισματικής αρχής. Είναι κάτι που το είχα θίξει και πέρυσι. Το ίδιο πλέον πρέπει να ελέγξουμε και τον ESM, ο οποίος είναι μηχανισμός ο οποίος δίνει ε, δάνεια στα κράτη-μέλη και μέσω του ESM εφαρμόζονται μνημόνια στα κράτη που λαμβάνουν τις, ε, τη δανειοδότηση. Άρα λοιπόν αυτά τα θέματα θεωρώ ότι είναι σημαντικά και θα τα θίξω στην, ε, στην έκθεσή μου. Επίσης σημαντικά είναι το θέμα του lobbying, το οποίο πρέπει να δούμε. Ο έλεγχος της Frontex στα θέματα των, ε, των δικαιωμάτων των, ε, των προσφύγων. Το δικαίωμα των καταγγελόντων, που επίσης είναι ένα σοβαρό ζήτημα και ε, επίσης το revolving doors, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό σε σχέση με το τι γίνεται με όσους ήταν στην Κομισιόν και μετά αν έχουν αναλάβει θέση. Άρα λοιπόν έτσι όπως παρουσιάστηκε η έκθεση από την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, νομίζω ότι είναι ε, μια πάρα πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει. Αυτές είναι πρώτες σκέψεις από πλευράς μου ως εισηγητή. Θα αναμείνω τους συναδέλφους, τους άντο ραπορτέρες για τις απόψεις τους. Αυτές είναι οι πρώτες σκέψεις για τα θέματα στα οποία μπορούμε να επικεντρωθούμε, ε, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλα ζητήματα που θα θίξουν οι συνάδελφοι και τα οποία θα προσπαθήσουμε να τα εντάξουμε στην έκθεσή μας που σε ένα μήνα περίπου θα καταθέσουμε εντός της προθεσμίας για να τη δουν οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά όταν, όταν μιλάτε για το, για το Eurogroup, ξέρουμε ότι θα γίνει πάρα πολύ, πολλά λόγια από εσά. Τώρα ήταν ενδιαφέρον, ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, η κυρία Πιτέρα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχά να συγχαρώ την κυρία Διαμεσολαβήτρια για την παρουσίαση που μας έκανε, η οποία ήταν πολύ πλήρης. Παρότι ήταν ευσύνοπτη, ήταν πλήρης. Μας παρουσίασε τα πιο σημαντικά θέματα που μας ενδιαφέρουν όλους και που που είναι πολύ σημαντικά για όλους όσους θέλουν να λειτουργούν σωστά τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε κάποια στοιχεία τώρα. Καταρχάς, μεγάλη πρόσβαση, έχουμε μεγάλη πρόσβαση στο και άνετη και απρόσκοπτη στο γραφείο σας. Ακούω πάρα πολλά θετικά σχόλια. Ακούω ότι το γραφείο του διαμεσολαβητή είναι πάντα ανοιχτό σε όσους έχουν ανάγκη, σε όσους θέλουν να προσφύγουν σε αυτό σε όλους όσους ενδιαφέρονται για την καλή λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Εγώ εδώ και πολλά χρόνια ενδιαφέρομαι για διοντολογικά θέματα και για θέματα διαφάνειας. Γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι πραγματικά για αυτή την έφαση που δίδεται σε ορισμένε περιπτώσεις σε αυτές ας πούμε, τις ε, περιστρεφόμενες πόρτες, ε, στα revolving doors ας πούμε, ε, θέματα τα οποία είναι πολύ επίμαχα θέλουμε να αποφύγουμε τέτοιες καταστάσεις. Είναι πολύ προβληματικές αυτές για ανθρώπους ε, όπως ας πούμε ευρωϊπάλληλοι που θέλουν να φύγουν από την ε, ευρωπαϊκή υπαλληλία ας πούμε και θέλουν να πάνε στο ιδιωτικό τομέα για να αναλάβουν άλλα καθήκοντα ας πούμε. Ε, αλλά που το κάνουμε με έναν τρόπο που υποσκάπτεται η εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι λοιπόν πολύ ικανοποιημένος για την, η κυρία πολύ ικανοποιημένη συγγνώμη, για αυτή την πρώτη έκθεση ε, που μας παρουσιάσατε. Εμείς όμως ως Ευρωβουλευτές θα πρέπει να επιμείνουμε στο εξή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταπολεμήσει πιο στεναρά αυτό το φαινόμενο των περιστρεφόμενων θυρών. Δεύτερο θέμα. Πολύ σημαντικό, εδώ και πολλά χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το θέμα της διαφάνειας των δραστηριοτήτων των ανθρώπων που ασχολούνται με τα λόμπι, που προέρχονται από τα λόμπι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ και χρόνια μα συνοδεύει ή φυστάμεθα λόμπι, α πούμε, και συνδέεται άρρηκτα με τη λειτουργία της πολιτική ζωής και, το, και με τη ζωή των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Προφανώς και θα πρέπει να έρθουν σε επαφή λομπίστε με του πολιτικού, με του βουλευτέ κτλ. για να του επηρεάσουν για να δώσουν και καλές, τους δώσουν και καλές ιδέες και να καταλήξουμε σε καλές νομοθετικές αποφάσεις. Αλλά δεν γίνεται πάντα με σωστό τρόπο και αυτό θέλω να τονιστεί στην εκθεσή μας. Θα ήθελα ακόμα μια φορά γενικά να συγχαρώ την διαμεσολαβήτρια. Νομίζω ότι η δουλειά που κάνει είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα και νομίζω ότι θα πρέπει να επωφεληθούμε από τη δουλειά του διαμεσολαβητή, γιατί νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες και πολύ ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Η Σολεδάδ. Σολεδάδ, το λόγο. Ευχαριστώ, Σεφίλια. Ευχαριστώ τη διαμεσολαβήτρια. Και εγώ θέλω να συγχαρώ με τη σειρά μου τη διαμεσολαβήτρια μετά από τα συγχαρητήρια που άκουσε από τους προηγούμενους συναδέλφους γιατί μας παρουσιάσει μια θαυμάσια δουλειά ε, όπως αυτή που έγινε μέσα στο 2015. Ε, επικεντρώθηκε στα πιο σημαντικά, στα πιο ενδιαφέροντα θέματα όπως το θέμα πούμε, της διαφάνειας που είναι μεγάλο μέλημα για τους πολίτες. Επίσης η ανάλυση του, της ε, διαφάνειας είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα να γίνει μια ανάλυση για αυτό το, θέμα. Επίσης, μπορεί να υπάρχουν πιθανές συγκρούσεις ε, μεταξύ διαφόρων φορέων. Ε, είναι πολύ σημαντικό το γραφείο της να αναλύσει αν ε, εξασφαλίζεται η η αποφυγή συγκρούσεων ε, συμφερόντων και εξασφαλίζεται και η ανεξαρτησία. Επίση, είναι τεράστιο πρόβλημα οι περιστρεφόμενε θύρε. Θα πρέπει να το αναλύσουμε αυτό το πρόβλημα. Και αν οι ρυθμίσει που έχουμε επαρκούν. Ε, όχι μόνο γιατί μπορεί να υπάρχουν συγκρούσει συμφερόντων ή διάφοροι πυρογνώμε που συμμετέχουν σε διάφορε επιτροπέ, α πούμε, αλλά θα πρέπει να δούμε αν η χρηματοδότηση αυτή τη υπηρεσία μα επιτρέπει να εξασφαλίσουμε την, το διαχωρισμό ανάμεσα στα ιδιωτικά συμφέροντα και τα δημόσια συμφέροντα και να εξασφαλίσουμε την πρωτοκαθεδρία του δημοσίου συμφέροντος. Συχνά ε, εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση και με ιδιωτικά κονδύλια. Μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι παρόλα αυτά έχουμε την επαρκή ανεξαρτησία. Επίσης, ε, να εφαρμόσουμε την σύμβαση του ΟΗΕ για τα άτομα με ειδικέ ανάγκες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και αυτό το θέμα και να τονίσω επίσης το θέμα των ψυχοσωματικών ασθενειών, ε, φυσικών, ε, είναι πολύ σημαντικό οι φυσικές ε, ασθένειες, αλλά και οι ψυχοσωματικές. Ορισμένα άτομα, ας πούμε, ε, έχουν ειδικά προβλήματα και άρα δεν έχουν το ίδιο στάτους με τα υπόλοιπα άτομα έναντι του νόμου, ας πούμε, λόγω της ε, ψυχικής τους κατάστασης. Ε, δικαίωμα ψήφου, παραδείγματος χάρη, το, ε, το δικαίωμα ψήφου περιορίζεται για τα άτομα αυτά σε πολλά κράτη-μέλη. Είναι τεράστιο θέμα. Αυτό πρέπει να τα δούμε όλα αυτά. Αυτή είναι μια πρόταση δική μου. Πρέπει να αναλύσουμε το πώς ε, εξασφαλίζονται αυτά τα δικαιώματα ε, των ατόμων αυτών και τα δικαιώματα επίσης των παιδιών. Συχνά τα παιδιά δεν έχουν φωνή. Θα πρέπει να βρούμε ένα μηχανισμό ώστε τα παιδιά να μπορούν να συμμετάσχουν ε, στη ζωή των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Για να δω πρέπει να αναλύσουμε πώς μπορούμε να το λύσουμε. Αυτά και τίποτε άλλο. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι εκφράσω και εγώ την ε, ικανοποίησή μου από τη δουλειά της διαμεσολαβήτριας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ σε φίλια. Και εγώ να συγχαρώ για την έκθεση αυτή. Μας δίνει ε, απίστευτα πολλές πληροφορίες, πολύ χρήσιμες. Επίσης, να σε συγχαρώ για τον τρόπο με τον οποίο ε, έκανες αυτή την έρευνα των, για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων της Κομισιόν. Υπάρχει μία ερώτηση ε, όπου αναφέρεται ότι θα πρέπει να γίνεται ένας ανοιχτός και δημόσιος διαγωνισμός για να επιλέγονται αυτοί οι εμπειρογνώμονες. Θα πρέπει να μας απαντήσει η Κομισιόν. Ε, όμως οι περισσότερες, ε, τα περισσότερα προβλήματα και παράπονα ε, ακούγονται λόγω της έλλειψης ε, διαφάνειας της εργασία της Κομισιόν. Αυτό δείχνει πολλά. Παραδείγματο χάρη, ε, αδιαφανείς είναι ε, πολλές σημαντικές διαπραγματεύσεις σε διεθνές επίπεδο. Το TTIP, το SETA κτλ. που γίνεται ε, χωρίς να ξέρει τίποτα ο πολίτης. Νομίζω ότι πορεύεται με επικίνδυνο τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση και οικοδομείται από πάνω προς τα κάτω και προωθεί πολύ συχνά ε, τα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά συμφέροντα, ε, τα συμφέροντα του κεφαλαίου και αυτό είναι ε, κάτι που απασχολεί τους πολίτες. Όπως είπε και άλλη Ισπανίδα συνάδελφος. Επίσης το, το δικαίωμα ψήφου είναι συχνά έρχεται σε αντίφαση αυτό το δικαίωμα ψήφου με το δικαίωμα στην κινητικότητα, ας πούμε. Σαν να ε, αντιπαρατίθεται το ένα απέναντι στο άλλο. Εάν έχεις δικαίωμα να εργαστείς σε οποιοδήποτε κράτο μέλο, είναι προφανές ότι θα πρέπει να ψηφίσει εκεί όπου εργάζεσαι και να μπορεί να ψηφίσεις από οποιοδήποτε κράτο μέλο. Δεν, να σου, δεν πρέπει να σου περιορίζουν το δικαίωμα. Επίσης υπάρχει πρόβλημα αδιαφάνειας λόγω αυτών των περιστρεφόμενων θυρών. Ε, το ξέρουμε αυτό το πρόβλημα στην Ισπανία. Και γιατί δεν δημοσιεύουμε πιο τακτικά τα ονόματα των ανθρώπων τα οποία φεύγουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πηγαίνουν σε άλλες δουλειέ, ας πούμε. Και αναλαμβάνουν άλλα καθήκοντα. Επίσης θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις. Μία. Τι απάντηση θα δώσει η Κομισιόν στι πρωτοβουλίε των Ευρωπαίων πολιτών όπω την πρωτοβουλία για το δικαίωμα σε πόσιμο νερό η Κομισιόν πάντα θα πρέπει να δίνει απάντηση σε ε, πρωτοβουλίες που συγκεντρώνουν τις απαραίτητες υπογραφές. Έτσι, τελειώνω, Σεσίλια. Θα πρέπει να απαντάει, λοιπόν. Έχετε λάβει α, παράπονα από τα μέλη που υποστήριξαν αυτή την πρωτοβουλία για τις απαντήσεις που δίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παραπονέθηκαν, λοιπόν, οι υπογράφοντες. Επίσης υπάρχει μια, ένα ψήφισμα του Ιουνίου του Κοινοβουλίου που ζητάει από την Κομισιόν να υπάρχει ένας κανόνας ε, διοικητική ε, διαδικασίας. Τι συνέπειες θα υπάρξουν αν υπάρχει ενιαία αυτή διαδικασία. Δεν, δεν θεωρείτε επίσης ότι αυτό δημιουργεί ανισότητες μεταξύ των πολιτών. Δίνω το λόγο στη Καλά, αγγλικά θα μιλήσω. Ε, έλεγα να μιλήσω δανέζικα, καλά δεν πειράζει. Καταρχάς, Έμιλη, να ε, σας ευχαριστήσω για τη δουλειά σας. Νομίζω ότι η Επιτροπή μας ε, μπορεί να είναι περήφανη που έχουμε πραγματικό διαμεσολαβητή. Νομίζω ότι ανταποκρίνεσαι στις προσδοκίες μας. Σε συγχαρητήρια λοιπόν. Δύο παρατηρήσεις. Να τονίσω καταρχάς ε, αυτό που είπαν αρκετοί συνάδελφοι όσον αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων. Εάν ε, εισάγουμε στη διοίκηση την αρχή της υπηρεσίας, η οποία σημαίνει ότι επικεντρωνόμαστε στους πολίτες, εξυπηρετούμε τους πολίτες, ε, ότι η διοίκηση δεν προστατεύει τους υπαλλήλους της. Έτσι θα έχουμε καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες και θα έχουμε ένα αξιοπρεπές και διαφανές ε, σύστημα. Και έτσι δεν θα υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Ε, μερικές φορές ο κόσμος ε, μπερδεύεται. Το ότι έχει κάνει κανείς δήλωση συμφερόντων δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Στο σύστημά μας, στη διοίκησή μας, ε, δεν επιτρέπεται να υπάρχει καθόλου. Για παράδειγμα, αν ακούσω ότι ε, κάποιος από τη φαρμακευτική βιομηχανία είναι σύμβουλος ε, της, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, δεν αρκεί αυτό. Θα πρέπει να γνωρίζω. Είναι αξιοπρεπής άνθρωπος, πληρώνει τους ε, φόρους του, είναι πιστός σε σύζυγό του. Ε, ε, αυτά μπορεί να μην με αφορούν, αλλά δεν θέλουμε καθόλου ανθρώπους με ε, σύγκρουση συμφερόντων που να λαμβάνουν τις αποφάσεις στο όνομα του συστήματος. Γι' αυτό υπάρχουν πολλοί τομείς όπου γίνεται πολύ καλή δουλειά και όσον αφορά τις περιστρεφόμενες πόρτες αλλά θα πρέπει να τονίσουμε ότι θα πρέπει ε, οι διοικήσεις μας για να είναι ε, αξιόπιστες ε, δεν θα πρέπει να επιτρέπουν καθόλου σύγκρουση συμφερόντων. Πώς το βλέπεις αυτό, διότι βέβαια δεν μπορούμε να προχωρήσουμε πέρα από τον νόμο, αλλά μπορούμε να απαιτήσουμε καλή τήρηση του νόμου. Και με τη συνθήκη λάβαμε μια υπόσχεση καλύτερης νομοθεσίας και βελτίωσης, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω δεν έχει γίνει τίποτα από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεύτερον, θα ήθελα να τονίσω, διότι αυτό μπορεί να φανεί πολύ σημαντικό σύντομα. Είσαστε η μόνη διαμεσολαβήτρια στον κόσμο με δικαίωμα να ε, ε, επικρίνετε το κοινοβούλιο σας, ε, εμάς δηλαδή. Και το δικαίωμα αυτό είναι υποχρέωση. Αυτά συνδέονται πολύ στενά στη δουλειά σας. Και δεν θα μπω σε συγκεκριμένες υποθέσεις, ε, αλλά νομίζω ότι διάφοροι από εμά έχουν διάφορες ιδέες σχετικά με το ποια θέματα θα πρέπει να επιβλέψεις εντός του Κοινοβουλίου, να εξετάσεις, να διερευνήσεις. Αλλά από ό,τι γνωρίζω, κανένας άλλος διαμεσολαβητής στον κόσμο έχει τέτοια δικαιώματα. Όχι στη Δανία, όχι αλλού από ό,τι ξέρω. Η δυνατότητα αυτή όμως συνεπάγεται και υποχρέωση. Και αν προσληθεί κανείς, μάλλον δεν έχει καταλάβει τι δουλειά κάνετε. Αλλά θα ήθελα πολύ ε, να σχολιάσετε αυτό το δικαίωμα, Παύλα, υποχρέωση. Ευχαριστώ πολύ. Η Ελεονόρα Εύη. Μάλιστα. Πολύ σύντομα θα πάρω, πολύ θα, σύντομα θα, θα πάρω το λόγο. Να μην επαναλάβω τα όσα είπαν οι συνάδελφοι που είναι αρκετά πλήρη. Χαίρομαι για την έκθεση που παρουσιάστηκε από εσά. Είμαι πεπισμένη ότι η δουλειά σας είναι θεμελιώδης για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, να τονίσω και ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν ε, ακούστηκε καθόλου, το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναφερθεί. Και είναι το θέμα της διαφάνειας στα μεγάλα δημόσια έργα και οι δυσκολίες που υπάρχουν και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τους Ευρωβουλευτές να πάρουν πληροφορίες, πραγματικές πληροφορίες, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση στα μεγάλα έργα, ας πούμε, τα οποία υλοποιούνται στην Ευρώπη γενικά. Ειδικά τα διασυνοριακά μεγάλα έργα. Ειδικά, ας πούμε, ε, η μεγάλη συνδρομική γραμμή Λιών-Τωρίνου. Εδώ και 20 χρόνια ξεκίνησε αυτό το έργο. Και είναι εντελώς περιττό, ας πούμε, έργο θα πρέπει να έχουμε περισσότερες πληροφορίες, μεγαλύτερη διαφάνεια, μεγαλύτερη πρόσβαση σε τεκμηρίωση. Και εμείς αλλά και οι πολίτες. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να αναφερθεί σε αυτή τη θαυμάσια έκθεση. Ήθελα να τονίσω λοιπόν αυτό το συγκεκριμένο στοιχείο που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ λοιπόν ακόμα μια φορά για τη δουλειά που κάνατε. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στο Γιάρεκ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, κυρία Ράιλι, είναι πάντα χαρά μας ε, να είσαστε εδώ μαζί μας. Ε, είναι εξαιρετική η δουλειά που κάνετε και χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ σήμερα στο βήμα. Κάτι που προσέλκυσε την προσοχή μου αναφέρθηκε ήδη ε, κάμια δυο φορές. Τον Γενάρη στείλατε επιστολή στην Επιτροπή ε, σχετικά με την ισορροπία όσον αφορά την επιλογή ε, πυρογνωμόνων και η Επιτροπή απάντησε ότι ναι, θα είναι πιο διαφανής η διαδικασία αυτή και καλέσατε την Επιτροπή να ε, δημοσιεύει τα αναλυτικά πρακτικά των ε, συναντήσεων των εμπειρογνωμόνων. Ε, εγώ εργάζομαι και στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και κατά τη γνώμη μου η διαφάνεια όσον αφορά τα λόμπι είναι απαραίτητη. Να σας δώσω παραδείγματα. Υπάρχουν ε, πολλές ε, διεθνείς οργανώσεις που εδρεύουν εδώ στις Βρυξέλλες και των οποίων οι απόψεις λαμβάνονται υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν εξετάσει κανείς όμως αυτές τις δίθεν ευρωπαϊκές οργανώσεις, διαπιστώνεται ότι μερικές από αυτές καθοδηγούνται από τρίτες χώρες ή παράγοντες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη έχω συζητήσει το θέμα με την κυρία Μάλμστρομ, δεν έχω λάβει όμως ε, θετική απάντηση, συγκεκριμένη απάντηση. Σας ερωτώ λοιπόν, ε, σκοπεύετε κι εσείς να εξετάσετε το θέμα αυτό, να διευρύνετε τις έρευνές σας πέρα δηλαδή από την διαφάνεια της επιλογής των εμπειρογνώμων και πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί τις απόψεις αυτών των δίθεν ευρωπαϊκών οργανώσεων στην νομοθετική της εργασία. Αγαπητοί συνάδελφοι, κλείσαμε τον κατάλογο των ομιλητών. Και δίνω πάλι το λόγο στην κυρία Οράιλη για να απαντήσει και να κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους που επένεσαν το έργο που επιτελούμε. Είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό και για το θεσμικό μας όργανο και για τους συναδέλφους στο θεσμό μας να έχουμε την υποστήριξή σας και ενδυναμώνεται για μας με αυτόν τον τρόπο η άποψή μας ότι βρισκόμαστε στη σωστή πορεία για θέματα ερευνών και προσπάθειες που μπορούν να καταλήξουν σε σχέση με το Κοινοβούλιο να είμαστε σε πολύ θετική σχέση. Καμιά φορά είναι πολύ μεγάλη πρόκληση για μας και για τα θεσμικά όργανα όλα αυτά και καμιά φορά είναι μοναχική δουλειά και είναι πολύ καλό όταν έχουμε ένα φόρουμ σαν εσάς και ε, βλέπουμε ότι συμμετέχετε όλοι μέσα σε ένα συνενετικό πλαίσιο και μας υποστηρίζετε. Για τα σχόλια και τις ερωτήσεις που έγιναν, κύριε Μωράης. Κύριε ε, Μαριά, ναι, το βιβλίο σας το έχω στο γραφείο μου. Και διαβάζω και ξαναδιαβάζω αυτά τα εδάφια, ιδιαίτερα όσον αφορά την παρέμβασή σας για το έργο που έγινε για παραβιάσεις. Ε, ε, μου θυμίζει το δικό μου έργο ότι πρέπει να έχουμε μακρόπνοη προσπάθεια σε σχέση με το, την ανταπόκριση που μπορεί να επιτευχθεί είναι πολύ σημαντικό και σε σχέση με το φόρουμ αυτό και για την Τρόικα και για θέματα δικαιωμάτων του ανθρώπου και για το πώς ε, άτομα και σε συγκεκριμένα καθεστώτα όπως και στην Ιρλανδία υπήρξαν συνθήκες όπου οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να υποστούν διάφορα δεινά. Και τώρα σε σχέση με το ότι μπορούν να, δουν το ότι μπορεί να λειτουργήσει το θέμα αυτό ξανά η Τρόικα και όλα αυτά θα πρέπει να τα ξαναδούμε και σε σχέση με το τι μπορώ εγώ να πράξω είναι σημαντικό το θέμα της διαφάνειας και να μπορέσουμε σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το, την Ευρωομάδα Eurogroup να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Και πάλι είναι επικοδομητικό αν έχουμε την υποστήριξη την δική σας. Εσάς ε, σας ευχαριστώ για τα σχόλια και για την ε, ε, της ε, δράσης ε, της, του θεσμού μας. Καμιά φορά είναι η τελευταία ίστατη λύση για, πολίτες που αισθάνονται απογοητευμένοι πολλές φορές και προσπαθούν να διασφαλίσουν τα δικαιώματά τους. Και προσπαθούμε, αν είναι δυνατόν, να ανταποκριθούμε στα αιτήματά τους. Συμφωνώ μαζί σας σε σχέση με το θέμα των περιστρεφόμενων θυρών και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν γίνεται λόγος για το δικαίωμα ανθρώπων να εργάζονται και πολλές φορές όταν ήταν στο ανώτατο επίπεδο κάποιοι που απασχολήθηκαν και όταν αποχωρούν και γίνονται προσφορές θελκτικές ε, για να εργαστούν αλλού, σίγουρα δεν είναι μόνο ένα θέμα ηθικής, είναι ένα θέμα ε, επιχειρηματικό για το πώς μπορούν να εργάζονται εκτός θεσμικών οργάνων άτομα που έχουν εκ των έσω τις πληροφορίες των δικών τους θεσμικών οργάνων. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει, αλλά και την ηθική υποχρέωση να είναι ο πυλωρός, ο θεματοφύλακας αυτών, ώστε αυτά τα οποία γίνονται να συνάδουν με το δημόσιο συμφέρον που πρέπει να διασφαλίζεται από την Επιτροπή και για το, τους λομπιίστες επίσης και η διαφάνεια από πλευράς λομπιιστών που πρέπει να διασφαλίζεται και σε σχέση με κάποιον από την Volkswagen και τις ε, πληροφορίες που πήραμε σε σχέση με τους περισσότερους που μπορεί να μην έχουν έναν άμεσο ρόλο σε αυτό. Είναι ένα θέμα όμως από την άλλη πλευρά ε, δικαιωμάτων του ανθρώπου. Όταν πρέπει να όταν έχουμε θέματα νομοθεσίας που έχουν επίπτωση στη ζωή όλων μας, έχουν δικαίωμα οι πολίτες να γνωρίζουν Πώς ε, καταρτίζονται αυτοί οι νόμοι, ποιες επιπτώσεις έχουν. Φυσικά εντάξει υπάρχει το δικαίωμα να δραστηριοποιούνται κάποιες λομπιίστες, αλλά πάλι πρέπει να διασφαλίζεται ένα πλαίσιο διαφάνειας. Συμφωνώ μαζί σας όσον αφορά τις ε, υπηρεσίες και τους οργανισμούς και πρέπει να εξετάσουμε και το θέμα του ότι ε, διασφαλίζεται πολύ σημαντικό έργο και όσον αφορά τα τα φάρμακα και την ε, συμβατότητά τους είναι όλο και πιο σημαντικά με την πάροδο των ετών και σε σχέση και με ε, κάποιον πανεπιστημιακό που ε, διορίζεται ως πραγματογνώμων ακόμα και σε ε, πλαίσια πιο εμπορικής δραστηριότητας είναι πολύ πιο δύσκολο να βρει κανείς καθαρά αυθεντικά ανεξάρτητους πραγματογνώμονες. Πρέπει όμως παρόλα αυτά να είμαστε αυστηροί σε σχέση με τα θέματα ηθικής για τα άτομα με ειδικέ ανάγκες, με μειονεξίες, πάρα πολύ σημαντικό θέμα αντιμετωπίζουμε παράπονα τα οποία έχουν ε, υποβληθεί από άτομα που εργάζονται σε θεσμικά όργανα και που έχουν παιδιά με ε, ειδικέ ανάγκες και πρέπει να γίνεται πάντα η προσπάθεια να διασφαλίζονται τα δικαιώματα αυτών των ατόμων υπάρχει και ένα δίκτυο, ευρωπαϊκό δίκτυο σε σχέση με τα παιδιά αυτά που έχει την έδρα του στο Στρασβούργο. Είναι σημαντικό αυτό το έργο να, το να αποτελέσει αντικείμενο που θα βοηθήσει στις εργασίες μας. Σε σχέση με τις προσπάθειες που έχουν γίνει, ε, γίνεται αντιληπτό ότι θα πρέπει σε σχέση με τα θέματα αυτά και την εμπιστοσύνη των πολιτών να ε, επιτηρούμε τα θέματα όπως πρέπει στην κυρία Άουκεν. Πράγματι, το Κοινοβούλιο εντάσσεται στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων μας και έχουμε και παράπονα τα οποία μας απασχόλησαν σε σχέση με το Ευρωκοινοβούλιο για την έκθεση και με τον τρόπο που αντιμετώπισε το Ευρωκοινοβούλιο άτομα που είχαν παιδιά με ειδικέ ανάγκες και που αυτό έθεσε, δημιούργησε μεγάλες πιέσεις και ένταση στις οικογένειες. <clears throat> σε σχέση με το Κοινοβούλιο δεν είναι πολύ εύκολο να ε, τραβηχτούν διαχωριστικές γραμμές. Είναι όμως μια υποχρέωση που οπωσδήποτε σέβομαι, ενώ από την άλλη μεριά θέλω να διασφαλίζω την ανεξαρτησία μου ως διαμεσολαβήτριας. Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα αυτών των θεμάτων, αλλά και την σπουδαιότητα του έργου των τριμερών διαλόγων και σε σχέση με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως και τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου έχω αποστείλει επιστολές ε, και για την ε, προώθηση αυτών των θεμάτων από πλευράς αυτών των θεσμικών οργάνων. Το κόστος ε, των πρωτοβουλειών αυτών, πολύ σημαντική υπόθεση, είναι σημαντικό για μένα τα παράπονα αυτά να μπορούν να μας οδηγήσουν στο να αντιμετωπίσουμε με ιδιαίτερη ευαισθησία αυτά τα θέματα. Σε σχέση με τα κράτη-μέλη, αν υπάρχει κάποια εμπλοκή σε σχέση με ε, συμβάσεις ε, ή τέτοιου είδους ε, υποχρεώσεις, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε, το οποίο θα μπορούσαμε να επιληφθούμε. Και μπορούμε σε σχέση με αυτό να συνδράμουμε. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ για τα πολύ θετικά σας σχόλια. Οι ομάδες πραγματογνωμόνων αυτό που αποφασίσαμε να πράξουμε είναι από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, έγιναν δεκτές κάποιες συστάσεις μας ε, όσον αφορά την ε, εφαρμογή τέτοιου είδους πρωτοβουλειών. Τελικά πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια και να υπάρχει μέσω ενός μητρώου η δράση που θα μας βοηθήσει να γνωρίζουμε για τη δραστηριότητα ατόμων που ασχολούνται σε συγκεκριμένους τομείς. Μία από τις επικρίσεις σε σχέση με τη διαφάνεια που διατυπώθηκαν είναι ότι δεν έχουμε αρκετά, αρκετές πληροφορίες για την χρηματοδότηση κάποιων ομάδων, ποιοι βρίσκονται πίσω από κάποιους συλλόγους και ενώσεις, όμως σε σχέση με την Επιτροπή Προϋπολογισμών και τις ε, δικές μας δράσεις ε, σε σχέση με αυτή την έκθεση και την ε, δράση των πραγματογνωμόνων ολοκληρώνοντας το έργο μας ολοκληρώνουμε αυτό το σκέλος σε σχέση με την διαφάνεια και νομίζω ότι αυτό αναπόφευκτα οδηγεί στο να διασφαλίζεται στο τέλος τέλος μεγαλύτερη διαφάνεια. Είναι σημαντικό αν υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις και ιδέες όπως από πλευρά σας για παράδειγμα να μπορείτε να προσέλθετε σε μένα να μου τις ε, γνωστοποιήσετε η, το θέμα της πληροφόρησης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να αποφύγουμε την παραπληροφόρηση και για το πόσο ε, ενεργά έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγγράψει αυτό το θέμα στις δραστηριότητές της. Και μέσω Google ή μέσω άλλης συλλογής στοιχείων σημαντικό είναι να γνωρίζει κανείς συγκεκριμένα για ποιο πράγμα γίνεται λόγος. Το να γίνεται λόγος για καλύτερη νομοθεσία είναι ένα πράγμα. Αλλά το να είμαστε πραγματικά εκεί που πρέπει αποτελεσματικοί είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι κάποια επανάσταση, αλλά είναι μια μετεξέλιξη. Είναι ένα θέμα εξέλιξης που βελτιώνεται εξελισσόμενο. Και όλο και περισσότερο, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση να διασφαλίζεται διαφάνεια. Το να αρνηθεί κανείς την διαφάνεια δεν είναι άρνηση μόνο έναντι των πολιτών μας, αλλά είναι και επιζήμιο στα ίδια τα θεσμικά όργανα. Και για το ίδιο το ευρωπαϊκό εγχείρημα <clears throat> αποβαίνει επιζήμιο Πρέπει να δημιουργείται ένα κλίμα εμπιστοσύνης σε σχέση με τους πολίτες και τα όσα τεκταίνονται από εμάς, από τα θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Οράγλη. Είναι προνόμιο, είναι πάντα μια πρόκληση και είναι και μια περιπέτεια όταν έρχεστε εδώ στην Επιτροπή μας. Μας εμπνέετε να παρακολουθούμε το έργο σας και μας ε, εμπνέετε να ασχοληθούμε με τα καθήκοντά σας. Θέλουμε να το κάνουμε σε στενή συνεργασία μαζί σας. Ήταν πολύ ενδιαφέρον και μας ανέπνευσε η παρουσία σας και η ομιλία σας. Συνάδελφοι, η έκθεση του κυρίου Μαριάς θα εξεταστεί στις 8 Σεπτεμβρίου και η καταληκτική ημερομηνία για τροποποίηση, είναι 26 Σεπτεμβρίου. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή αρχές Νοεμβρίου και εν συνεχεία θα πάει στην Ολομέλεια στα τέλη του έτου. Θα δώσω το λόγο στους ε, αναφέροντες σε λίγα λεφτά. We, what we have to do because ο συντάκτης, ο, αναφέρον για την ε, υπαριθμόν 6 αναφορά ε, δεν έχει φτάσει ακόμα. Επομένως, προτείνω να περάσουμε στην ε, αναφορά 7, αριθμός 246 του Αλμπέρτο Τσίριο, με 15.000 υπογραφές για την κατασκευή μιας εγκατάστασης για την απόθεση φθαρμένων ελαστικών στο Ρετορμπίντο στην Ιταλία. Θεωρήθηκε παραδεκτή αυτή η αναφορά με βάση τη διαδικασία κατεπήγοντος, γιατί αφορά την έγκριση για την κατασκευή ε, ενός, ε, μιας εγκατάστασης στη Λομβαρδία για την ε, απόθεση φερμένων ελαστικών. Οι περιφερειακές αρχές της Λομβαρδίας θα πάρουν απόφαση 31 31 Ιουνίου, εννοεί 30 Ιουνίου προφανώς συνεδρία η το δημοτικό Είχαμε λάβει λοιπόν κατεπίγουσα απόφαση να βάλουμε στη σημερινή μερίσια διάταξη αυτό το θέμα. Ε, καλωσορίζω την προσωπία από τη Βογγέρα. Είναι εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο, οι εκπρόσωποι από το Δημοτικό Συμβούλιο. Σας καλωσορίζω. Θα ήθελα να δώσω το λόγο καταρχήν στον κύριο Ευχαριστώ. Κύριο εννοεί η πρόεδρος φυσικά. Ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Σας ευχαριστώ που επιτρέψατε τη διαδικασία του, του κατεπήγοντος για να εξετάσουμε αυτή την αναφορά με αυτή τη διαδικασία. Γιατί μιλάμε για μια εγκατάσταση που η άδειά του ε, εξετάζεται από τις περιφερειακές αρχές και αντιμετωπίζαμε τον κίνδυνο, πραγματικό και απτό κίνδυνο, να γνωμοδοτήσουμε πάνω σε κάτι το οποίο έχει ήδη επιτραπεί να γίνει, έτσι. Άλλο, αλλά χάρη στη διαδικασία του κατεπήγοντος δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Μιλάμε λοιπόν για μια εγκατάσταση για την διάθεση φθαρμένων ελαστικών. Και μιλάμε για αυτή την κοινότητα του ρετόρντιντος στη Λομβαρδία, στην Ιταλία. Πίσω μου υπάρχει μια εκπροσώπηση με, βλέπετε με την Ιταλική σημαία και τα επίσημα ρούχα. Όλοι οι, οι κάτοικοι ήταν κατά της α, ε, δημιουργίας αυτής της εγκατάστασης. Γιατί εκφράζουν καταρχάς αμφιβολίες για την νομική πτυχή, δηλαδή για, την, για το κατά πόσον είναι σωστή η διαδικασία χορήγησης άδειας, αλλά και για το, πρέπει να, για το κατά πόσο θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο, μια τέτοια εγκατάσταση. Είμαστε στην ε, ε, Παιδιάδα του Πάδου, έτσι, στην κοιλάδα του Πάδου. Ε, επίσης έχουμε θέρμες εκεί πέρα. Είναι γνωστή αυτή η περιοχή. Ε, είναι και αγροτική περιοχή επίσης. Όλα αυτά ε, συγκλίνουν προς το ότι δεν θα έπρεπε να γίνει μια τέτοια εγκατάσταση εκεί. Τώρα, θα αφήσω το λόγο στον ε, δήμαρχο του Ρετόρντιντο. Ε, θα μας μιλήσει συνοπτικά, αλλά και πολύ συγκεκριμένα, ποια είναι τα προβλήματα σε σχέση με αυτή την εγκατάσταση. Να πω στους αδέλφους μόνο ότι σας ευχαριστώ βεβαίως για την κατεπίουσα διαδικασία. Ε, χρειαζόμαστε ε, να κοινοποιήσετε την απόφαση, όποια και αν είναι αυτή, στις Ιταλικές αρχές, έτσι. Ούτως ώστε να ακουστεί και η θέση της Ευρώπης ε, στην Ιταλία με ηχηρό τρόπο. Μετά από αυτά θα δώσω το λόγο στην Ιζαμπέλα Τσεμπρέλη, που είναι η δήμαρχος του Ρετόρμπιντο. Ευχαριστούμε την, την Επιτροπή και τον κύριο Τσίρια η εγκατάσταση αυτή ε, θα γίνει στην Επίτροπο ε, ε, Ρετόρμπιτο. Τον Ιούλιο του 2014 εκφράστηκε η διάθεση από μία εταιρεία να γίνει μία έκθεση για την περιβαλλοντική επίπτωση. Αυτή η ίδια η εταιρεία που ασχολείται και με την ενέργεια παρουσίαζε στην ε, περιφέρεια της Λομβαρδίας στην, Επιτρο... στην κοινότητα του Ρετόρπιτο ένα έργο για την ε, υλοποίηση ενός, ε, μιας εγκατάστασης ανακύκλωσης τέτοιων θαρμένων ελαστικών. Θα χρησιμοποιήσει μια τεχνολογία Ε, θερμικής επεξεργασίας με βάση την πυρόληση. Ο στόχος της εγκατάστασης είναι η 100% ανακύκλωση και ανάκτηση του, των υλικών από τα οποία αποτελείται αυτό το ελαστικό ή τα, ελαστικά. Ε, βαριά δηλαδή και ελαφριά ε, υδρο, υδρογονάρθακης, ε, μαύρος άνθρακας ε, κτλ. Ε, σε πειραματικό στάδιο αυτή η τεχνολογία υπάρχει μόνο στην Ιαπωνία. Δεν έχουμε τη δυνατότητα δηλαδή ε, να δούμε τι θα γίνει με, την, ε, με τις οσμές και με τις εκπομπές που θα εκλείονται στην ατμόσφαιρα. Επίσης, στην, ε, στο Καζαλίνο, στην επαρχία της Νοβάρας, αρνήθηκαν να φτιάξουν αυτή την εγκατάσταση. Αρνήθηκε δηλαδή η περιοχή αυτή. Η δική μας περιοχή τώρα είναι πάρα πολύ σημαντική υδροθερμική δεξαμενή. Επίσης υπάρχει μια πολύ προχωρημένη γεωργία που δίνει πολύ καλά ε, γαστρονομικά προϊόντα και αμπελοϊνικά προϊόντα. Αν εγκατασταθεί εκεί αυτή, αυτό το εργοστάσιο θα είχε τεράστιες επιπτώσεις και στον τουρισμό ε, και στις, ε, στα τρόφιμα που παράγονται ε, θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα στο περιβάλλον και στον τουρισμό ε, και θα έθετε να αμφιβόλω πολλές θέσεις απασχόλησης. Η κοινότητα του Ρετόρμπικο μαζί με την επαρχία της Παβίας την Λομβαρδία έχουν κάνει ε, πολύ μεγάλες επενδύσεις ε, για το Greenway, που είναι ένας ε, ποδηλατόδρομος που ξεκινάει από τη Βογγέρα και φτάνει στο Ρετόρμπιντο, περνώντας μέσα από διάφορες θέρμες και στο μέλλον προβλέπουμε να φτάσει μέχρι το Βάτσι, που είναι η, η Κομόπολη, που είναι πρωτεύουσα του, της επαρχίας του Τρεβίζα. Διατρέχουμε δηλαδή ουσιαστικά μια μεγάλη περιοχή που θα, όπου εκεί ακριβώς θα εγκατασταθεί ε, το εργοστάσιο πυρόλησης. Επίσης έχουμε πολλές εγκαταστάσεις, ε, πολλές εκμεταλλεύσεις αμπελοϊνικές. Κανείς μπορεί να κάνει με τα πόδια μια, μια υπέροχη διαδρομή ας πούμε και να γευτεί διάφορα προϊόντα, ε, κρασιά κτλ. Έχουμε την εταιρεία Ντόρνο που φτιάχνει πολύ ωραία κρασιά. Ε, στη Βογγέρα έχουμε μία άλλη ε, έτσι, εγκατάσταση και τα λοιπά και μια εταιρεία που φτιάχνουν ε, πολύ ωραία τρόφιμα ονομασίας προέλευσης. Εάν φτιάξουμε και το εργοστάσιο της πυρόλησης θα ήταν μια καταστροφή. Λίγα μέτρα από αυτή την περιοχή έχουμε και ένα χήμαρο, ένα χήμαρο ε, έχουμε επίσης πολύ κοντά ε, την περιοχή ε, που ζουν οι άνθρωποι, οι κάτοικοι ας πούμε. Έχουμε σχολεία, έχουμε οίκους ευγυρίας, έχουμε τις πολύ ωραίες θέρμες και επίσης έχουμε κοντά και ένα αεροδρόμιο. Αυτή η ζώνη είναι πολύ γνωστή. Είναι η είσοδος για να μπει κανείς στην κοιλάδα που βρίσκεται κοντά του πάντου. Είναι υπέροχη αυτή η κοιλάδα. Όπως είπαμε ήδη, είμαστε σε μια πολύ σημαντική υδροθερμική ε, δεξαμενή που είναι μοναδική περίπτωση στην Ιταλία. Ε, τα, νερά αυτά στις θέρμες έχουν, ε, περιέχουν και θείο και οι όδιο έχουν πολύ, πολύ μεγάλες και σημαντικές ιαματικές ιδιότητες, είναι γνωστές από την ρωμαϊκή εποχή και είναι γνωστές όχι μόνο στην περιοχή μας αλλά και εκτός, στην Ιταλία και εκτός. Ε, ξαναλειτουργήσαν οι θέρμες αυτές από την αρχαία εποχή από το 1860. Ε, ε, το 2009 ε, δημιουργήθηκε ένας νόμος για να ε, φτιάξουμε, να μεταφέρουμε τον τόπο των θερμών αυτών. Ε, ανοίξαμε μια, μια νέα εγκατάσταση δηλαδή. Ε, επίσης, αρχικά ε, το χωριό που ήταν η Θέρμες λεγόταν Κοντιάσκο. Τώρα λέγεται Κοντιάσκο Σάλιτσι Θέρμες. Με αυτές τις δράσεις η επαρχία της Παβίας και με την αλλαγή των ονομάτων ε, προσπαθεί να προωθήσει αυτές ε, τις θέρμες. Ε, δημιούργησε και αυτό το ποδηλατόδρομο και πεζόδρομο για να προωθήσει τουριστικά την περιοχή, να χρησιμοποιήσουμε την, τον πλούτο που έχει σε γαστρονομικό και αμπελονικό επίπεδο κτλ. Για όλα αυτά, για όλες αυτές τις προσπάθειες που έχουν γίνει, για όλες τις επενδύσεις, η περιοχή της Λομβαρδίας δεν θα πρέπει να επιτρέψει να εγκατασταθεί εκεί ένα εργοστάσιο πυρόλησης. Η εγκατάσταση αυτή, όπως σας είπαμε, θα δημιουργούσε ε, πολλά προβλήματα σε όλη αυτή τη ζώνη και θα ακύρωνε αυτές τις επενδύσεις. Θα θέλαμε να πούμε ότι το σχέδιο της κυβέρνησης ε, της ε, επαρχίας αυτής είχε πει ότι δεν θα πρέπει να δημιουργηθεί καμία εγκατάσταση κανένα εργοστάσιο το οποίο θα έχει, χρησιμοποιεί ε, επικίνδυνα υλικά, θα είναι επικίνδυνο για το περιβάλλον αυτό κτλ. Όπως ακριβώς η εγκατάσταση για την οποία μιλάμε. Επίσης, έχουμε στο Κόρτε Λεόν ε, μια εγκατάσταση αποτέφρωσης ε, που χρησιμοποιείται για να διαθέσουμε απορρίμματα. Επίσης, στο Σάντα Λαζάρο, την Μπορμπόνη, καζατίσμο Τσερβέζο, ε, Γκαμπολόνε, Ρέτο, ε, έχουμε ε, χωματερές που χρησιμοποιούν τσιμέντο και αμίαντο στο Κάβα Μανάρο. Επίση, έχουμε μια, ένα δηληστήριο το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, στη Βερένα Φερέρα Εμπορνιόνη και στο Σαλατζάρο την Μπορμπόνε. Έχουμε όμως εκεί ακριβώς λόγω αυτών των ε, εγκαταστάσεων ε, μόλυνση από αμίαντο. Έχουμε 15 εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ε, ορισμένα χρησιμοποιούν τη βιομάζα. Παρουσιάσαμε στον πρόεδρο της περιοχής της Λομβαρδίας, τον κύριο Μαρόνι, και στην σύμβουλο της περιοχής της Λομβαρδίας, τη Κλάουντια Τέρτσι, όλα τα προβλήματα και όλες τις αμφιβολίες, όλους τους φόβους των πολιτών της περιοχής μας. Είμαστε κατά της ε, εγκατάστασης. Έχουμε καταθέσει 130 υπογραφές των ε, δημάρχων και περίπου 100.000 υπογραφές από πολίτες. Ε, ζητάμε από τους αρμόδιους να σταματήσει η οικοδόμηση και εγκατάσταση αυτής της ε, εκμετάλλευσης. Σας ευχαριστώ που οργανώσατε αυτή την ακρόαση και που μας δώσατε τη δυνατότητα να παράγουμε το λόγο για να σας εξηγήσουμε τα προβλήματα που θεωρούμε ότι υπάρχουν. Ζητάμε από την Επιτροπή σας να εκφραστεί η θέληση των πολιτών της περιοχής της Παβίας, ε, η θέληση των ε, τοπικών και περιφερειακών αρχών, των δημάρχων κτλ. Και θα θέλαμε η Επιτροπή να μιλήσει στην, στις αρμόδιες Ιταλικές αρχές, ούτω ώστε να μην υλοποιηθεί αυτή η εγκατάσταση, που πέρα από τις περιβαλλοντικές καταστροφές, πέρα από τις καταστροφές στο τοπίο και στις οικονομικές καταστροφές, θα δημιουργούσε και τεράστια προβλήματα στην υγεία. Ελπίζουμε ότι όλα αυτά που σας είπαμε θα τα ακούσετε με βίκο νους και σας, χαιρετούμε, σας χαιρετίζουμε. Καλούμε επίσης την Επιτροπή μέσω του κυρίου Τσίριου να έρθει στο, στο, στην περιοχή μας, εκεί όπου θα εγκατασταθεί αυτή, αυτό το εργοστάσιο, ε, να γευτείτε τα κρασιά μας και τα τρόφιμά μας για να καταλάβετε τι παράγουμε. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Συνάδελφοι, λέγομαι Τσάκη. Μου ζητήθηκε από την Πρόεδρο, να αναλάβω την Προεδρία της Επιτροπής και να διευθύνω τον διάλογο για το θέμα αυτό. Θα μιλήσω σλοβάκικα, εάν μου το επιτρέπετε. Θα ήθελα να παρακαλέσω την κυρία Μανταλένα Καπούσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει το λόγο. Γενική Διεύθυνση ΕΝΒΗ. Καλό απόγευμα σε όλους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους ε, αναφέροντες που βρίσκονται σήμερα εδώ για να παρουσιάσουν τη θέση τους ε, που είναι κατά της ε, δημιουργίας μιας εγκατάστασης για την ανακύκλωση μεταχειρισμένων ελαστικών. λαμβάνουμε γνώση της αναφοράς και καθότι διαβιβάστηκε μόλις την τελευταία εβδομάδα το θέμα αυτό σε εμάς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόμα διαμορφώσει θέση πάνω στην αναφορά αυτή. Ωστόσο, όπως πάντα, ακούμε τις θέσεις και θα εξετάσουμε προσεκτικά την αναφορά αυτή και θα μεταφέρουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη θέση μας. Θα πούμε δηλαδή αν μπορούμε να βοηθήσουμε τον ε, αναφέροντα και τι δράση μπορεί να αναλυθεί από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επίτροπή όσον αφορά το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε καθυστερήσει. Τέσσερις συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Φυσικά θα τους δώσω χρόνο ομιλίας, ωστόσο θα ήθελα να είμαστε όλο πιο, όσο πιο σύντομοι γίνεται σε αυτήν τη συζήτηση. Προτείνω λοιπόν να παραμείνει σε κρεμότητα η αναφορά αυτή, διότι είναι σοβαρό το θέμα. Και δεύτερον, να περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τρίτον, ε, αυτή τη βδομάδα να στείλουμε επιστολή στις περιφερειακές αρχές σας στην οποία θα εξηγούμε τη δυσαρέσκειά μας ε, για το σχέδιο αυτό και θα ζητάμε περισσότερες πληροφορίες. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν καλό να γίνει. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Κυρία Καβεθό, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε σε σχέση με τα όσα αναφέρθηκαν από τον αναφερόμενο. Σε σχέση με την ίδια την ανησυχία μας για τις επιπτώσεις σε σχέση λοιπόν Ανησυχ... Ε, κατανοούμε πάρα πολύ για την ανησυχία σε σχέση με την εγκατάσταση αυτής της ε, μονάδας στην περιφέρειά τους. Όταν κάνουμε λόγο για την ανακυκλούμενη οικονομία και την ε, δυνατότητα της ε, απάλληψης ή άλλης χρήσης αυτών των αποβλήτων. Θα πρέπει να αναζητηθούν άλλες λοιπόν εναλλακτικέ λύσεις και αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η γνωμοδότηση σε σχέση με την Επιτροπή, τι θα πούν οι αρχές θα πρέπει να αναζητηθούν λοιπόν άλλες ε, πιο αποτελεσματικές δυνατότητες σε σχέση με την ε, ίδια αυτή περίπτωση με απόβλητα απολάστιχα είχαμε μια τεράστια πυρκαγιά στην Ισπανία και η κατάσταση ναι μεν ελέγχθηκε αλλά ε, η κατάσταση ήταν πάρα πολύ πιεστική η μόλυνση του ατμοσφαιρικού αέρα η πίεση όσον αφορά το περιβάλλον πρέπει να αναζητηθούν εναλλακτικέ λύσεις σε τέτοιου είδους απόβλητα και να είμαστε πιο αηφόροι όσον αφορά το περιβάλλον. Μαριάς παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στηρίξαμε και εμείς ως CCR τον ε, συνάδελφο από την Ιταλία, ο οποίος ζήτησε να υπάρξει μια διαδικασία κατεπήγοντος την εξέταση της αναφοράς. Και είναι πολύ σημαντικό, το υποστηρίξαμε και σήμερα νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας την δυνατότητα να πάρουμε μια πρώτη απόφαση. Διότι είναι ξεκάθαρο, το εξήγησε ο συνάδελφος Ευρωβουλευτής αλλά και η Δήμαρχος, ότι εδώ πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα οικολογικά στο περιβάλλον, στον τρόπο ανάπτυξης περιοχής, στην υγεία των κατοίκων, ιδίω όταν έχουμε ένα εργοστάσιο πυρόλησης. Άρα λοιπόν αυτό είναι δεδομένο. Από την άλλη γνωρίζαμε όταν συζητήσαμε στην, στους συντονιστές ότι πιθανόν η Κομισιόν, επειδή μόλις θα λάβει την, την ε, αναφορά, πιθανόν να μην μπορεί να έχει την δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις της. Επομένως, κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με την πρόταση που κάνατε, συμφωνούμε στα εξή. Πρώτον, να υπάρξει μια επιστολή πρώτα απ' όλα στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ιταλίας. Διότι εδώ είναι ένα θέμα σοβαρό, αφορά, όπως λένε οι καταγγέλλοντες, παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα του περιβάλλοντος και της προστασίας της δημόσιας υγείας. Επομένως η επιστολή πρέπει να πάει προς την μόνιμη αντιπροσωπεία της Ιταλίας. Δεύτερον, η επιστολή όπως είπατε πρέπει να πάει στις περιφερειακές αρχές οι οποίες είναι να λάβουν την απόφαση σε λίγες μέρες. Αλλά στην επιστολή προτείνω να τους ζητήσουμε όχι μόνο πληροφορίες αλλά να τους ζητήσουμε να μην λάβουν καμία απόφαση μέχρι ότου να έχουμε τη γνώμη της Κομισιόν. Δηλαδή να αναστείλουν κάθε απόφαση η οποία πρέπει να ληφθεί από τις περιφερειακές αρχές. Αυτό πρέπει να το πούμε ρητά στην επιστολή μας, ούτω ώστε να καταστήσουμε τις περιφερειακές αρχές υπεύθυνε. Εάν η Επιτροπή έρθει και γνωμοδοτήσει ότι πρόκειται για παραβίαση της νομοθεσίας, να θεμελιώνεται πλέον ευθύνη των περιφερειακών αρχών της Ιταλίας και βεβαίως της Ιταλικής πολιτείας για παραβίαση των δικαιωμάτων των ίδιων των πολιτών. Αυτό πρέπει να πούμε στην επιστολή μας και αν συμφωνούν οι συνάδελφοι αυτό είναι σημαντικό και ίσως πλέον κύριε Πρόεδρε και τελειώνω να είναι και ένα τεστ. Δηλαδή αν οι Ιταλικές Περιφερειακές Αρχές αναστείλουν τη λήψη απόφασης θα αποδειχθεί ότι η Επιτροπή μας είναι αποτελεσματική και σε τέτοιες έκτακτες περιπτώσεις και άλλες φορές θα μπορούμε να φέρνουμε αναφορές κατεπηγόντως να τις εξετάζουμε και να λύνουμε το πρόβλημα πριν δημιουργηθεί. Διότι αυτός είναι ο ρόλος μας. Άρα λοιπόν συμφωνώ με τις παρατηρήσεις σας, συμφωνώ με όσα είπαν οι συνάδελφοι και να προσθέσουμε αυτό το σημείο. Οι περιφερειακές αρχές της Ιταλίας να κληθούν να μην λάβουν καμία απόφαση μέχρι ότου να έχουμε τη γνώμη της Κομισιόν επί του ζητήματος που συζητούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Δαλιάνα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με την πρόταση που έγινε από σε Προέδρου και σε σχέση με την πρόταση του κυρίου Μαρία γιατί πρέπει να έχουμε την αρχή της προφύλαξης εδώ, της πρόνοιας σε σχέση με αρνητικότητες επιπτώσεις τέτοιων μέτρων ή πρωτοβουλειών για την ε, πυρόληση και την επιβάνηση του ατμοσφαιρικού αέρα και ξέρουμε επίσης ότι υπάρχει εδώ πολύ μεγάλος κίνδυνος μόλυνσης, ρήπανσης από τέτοιου είδους λάστιχα. Και ακριβώς στη χώρα μας μέχρι τις 2 Ιουνίου είχαμε σε μια παράνομη χωματερή μια τέτοια περίπτωση πυρκαλιάς, 100.000 τόνοι ελαστικών είχαν υποστεί αυτή την ε, ε, πυρκαλιά και όταν ε, άρχισε η αφαίρεση των ε, λαστικών εκείνων που δεν είχαν ε, πάρει φωτιά υπολογίζεται σε χιλιάδες τόνους αυτός ο όγκος και η κυβέρνηση της Καστίγια Λαμάτσα Αποφάσισε ότι πρέπει, ε, θα έπρεπε να δημιουργηθεί μια δυνατότητα ώστε να χρησιμοποιηθούν αυτά σε σχέση με ε, κτίρια. Ακόμα μεγαλύτερη δηλαδή περίπτωση ε, ρήπανσης. Πρέπει να αφήσουμε ανοιχτή αυτή τη δυνατότητα όπως προτάθηκε. Πρέπει να μάθουμε, να συναγάγουμε τα συμπεράσματα από αυτά που συνέβησαν στην Ισπανία και πρέπει να αποφύγουμε χειρότερα ακόμα τέτοια περιστατικά και να δώσουμε, να κάνουμε εκείνο το οποίο είναι αναγκαίο ώστε να αποφύγουμε τέτοιου είδου συμβάντα στο μέλλον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ τους δημάρχους που είναι παρόντες εδώ. Ευχαριστώ τις Ιταλικές αρχές και όλους όσους υποστήριξαν αυτή την αναφορά. Είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας να ταχθεί και να μιλήσει ξεκάθαρα για τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να γίνει αυτή η εγκατάσταση. Είναι μια παλιά, είναι ένα παλιό, μια παλιά τεχνολογία αυτή. Δεν έχει καμία σχέση με αυτά που θέλουμε σήμερα που είναι η κυκλική οικονομία. Και επιπλέον έχει συσσωρευτικές επιπτώσεις μαζί με όλες τις άλλες εγκαταστάσεις αποτέφρωσης που έχουμε ήδη κτλ. Ε, Όλα αυτά είναι πάρα πολύ αρνητικά, θα πρέπει να τα αποτρέψουμε. Να σας υπενθυμίσω κάτι. Έχουμε τον, το διγλιστήριο αυτό, έχουμε την ε, χωματερή αμίαντου, έχουμε τους αποτεφρωτές. Ε, έχουμε δηλαδή πολλές εγκαταστάσεις εκεί και όμως αυτή είναι μια πολύ σημαντική ε, γεωργική περιοχή αν φτιάξουμε και αυτήν την εγκατάσταση, θα έχουμε σωρευτικά αποτελέσματα. Επίσης, να υπενθυμίσω ότι στην ε, Επιτροπή μας μιλήσαμε για την ε, ποιότητα του αέρα και μιλώντας για αυτό το θέμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε ότι η Λομβαρδία θα μπορούσε να ξαναμπεί ε, να είναι σε παράβαση μάλλον και να υπάρξει προσφυγή της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της περιοχής της Λομβαρδίας λόγω του, του ότι υπάρχει πρόβλημα με την ποιότητα του αέρα. Ένας ακόμα λόγος για να αποφύγουμε την κατάσταση τέτοιων εργοστασίων που σε καμία περίπτωση δεν προστατεύουν ούτε την υγεία ούτε το περιβάλλον. Και όπως είπε και ο Νότης, ναι, πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτή την ε, αναφορά αυτή, να στείλουμε μια επιστολή πολύ γρήγορα στις Ιταλικές Αρχές Και σίγουρα όλα αυτά να τα συνδέσουμε και με απάντηση τη ε, Κομισιόν και να περιμένουμε σίγουρα απάντηση από την Κομισιόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τους ε, αναφέροντες και τον συνάδελφο Τσίριο για το ότι ε, ενεγράφει αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη απόψε και με σύμφωνη γνώμη των συντονιστών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό διότι έχουμε μια κατάσταση απέναντί μας όπου έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για αυτό το εγχείρημα και ξέρουμε ότι όταν έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι διαδικασίες είναι πολύ δύσκολο να υπάρξουν τροποποιήσεις, αλλαγές, ε, βελτιώσεις και είναι πάρα πολύ σημαντικό και να δούμε ότι στην ίδια τη διαδικασία πριν από την έγκριση να μπορούν να, γίνουν, να εισακουστούν τα επιχειρήματα των αναφερόντων γιατί διαφορετικά χρησιμοποιούμε πάντα το ρόλο του παθολόγου. Δηλαδή είναι άρρωστος ο ασθενής και πρέπει ο γιατρός να τον θεραπεύσει, ενώ μπορούσε να έχει προληφθεί η ασθένεια. Το ανέφερε καλά η πρόεδρος και εν τη ε, Σοφία της ε, ανέφερε ότι πρέπει να προπαρασκευαστούμε και να ζητήσουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρόμοια με τον, την ίδια ταχύτητα και με τον ίδιο έντονο τρόπο όπως ε, οι αδειοδοτούσες αρχές να μεριμνήσει διότι από πλευρά της Επιτροπής υπάρχουν υπεύθυνοι που θα πρέπει να αναφέρουν στους κρατικά υπεύθυνους ότι η κοινοτική νομοθεσία πρέπει να είναι σεβαστή και έχουμε την ε, οδηγία πλαίσιο ότι πρέπει να υπάρξει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και όλα αυτά θα πρέπει σε μια παράλληλη διαδικασία να αποτελέσει αντικείμενο αρρωγής ε, επικοδομητικά να μπορέσουμε να δράσουμε να δώσουμε τη μάχη σε ένα μέτωπο και τέταρτον πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά και σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις μας να μας ξανααπασχολήσει όταν θα έχουμε κάποιες απαντήσεις ή στοιχεία στα χέρια μας. One minute. Για ένα λεπτό, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, λέει ο Τσίριο, και να επαναλάβω, Πρόεδρε, πέρα από το γράμμα που θα στείλουμε για να δείξουμε ότι η Ευρώπη έχει τα μάτια στραμμένα εκεί, το βασικό είναι να, να σταματήσουμε και τη διαδικασία που είναι εν εξελίξη. Μέχρι να λάβουμε την επίσημη ε, άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν το καταφέρουμε αυτό θα είναι πολύ θετικό το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Συνοψίζω λοιπόν. Παραμένει ανοιχτή η αναφορά θα, στείλουμε, αναφορά, θα στείλουμε δύο επιστολές. Ένα στη μόνιμη Ιταλική Αντιπροσωπεία και ένα δεύτερο γράμμα στις ε, περιφερειακές αρχές όπως αναφέρατε. Και τρίτον, θα περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνείτε. Ευχαριστώ κύριε και κύριοι. Έχουμε τελευταία αναφορά σήμερα. Του 2015 υπαριθμών 1049. Έχουμε ένα Ιταλό αναφέροντα εδώ και το θέμα της αναφοράς είναι το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δυστυχώς, η αναφέρουσα δεν έχει φτάσει, παρότι την καλέσαμε στην συνεδρίαση αυτή. Θα ήθελα να ζητήσω αν η κυρία Ανεμοντάνιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ο κύριος Μάουερ μπορούν να πάρουν το λόγο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Υποβάλλω μια πρόταση, αλλά ανακοινώνεται από πλευρά του αναφέροντος ότι δεν είναι δυνατόν να προσέλθει. Δεν γνωρίζω αν είναι δυνατόν να ε, υπάρξει μια αλλαγή ώστε να εξεταστεί αυτό το θέμα σε άλλη συνεδρίαση της Επιτροπής. Γεια σας. Ο κύριος Λούτσο Λέβη δεν έχει καταστάσει ακόμα. Θα ήθελα όμως αν είναι δυνατόν να παρουσιάσω εγώ την αναφορά. Επιτρέψτε μου, νομίζω ότι αυτό είναι κάπως προβληματικό. Αλλά να ρωτήσω πρώτα τους εκπροσώπους της Επιτροπής ποια είναι η θέση τους. Κατόπιν ε, ίσως να έχετε τη δυνατότητα να παρέμβετε. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να κάνω κάποιες παρατηρήσεις από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πάνω σε αυτήν την αναφορά. Να σας παρουσιάσω το πλαίσιο, διότι υπάρχουν διάφορα θέματα που αναφέρονται στην αναφορά αυτή. Το πρώτο είναι η ενδιάμεση αναθεώρηση. Όπως γνωρίζετε, η ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιετούς ε, δημοσιονομικού πλαισίου θα μας δώσει μια ευκαιρία να εξετάσουμε πώς λειτουργεί το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και επίσης θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο τον προϋπολογισμό για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που δυστυχώς κληρονομήσαμε από την χρηματοοικονομική κρίση και ιδιαίτερα το κενό των επενδύσεων, την έλλειψη επενδύσεων. Και αυτό σχετίζεται με το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις Στρατηγικές Επενδύσεις ε, και τα ομόλογα έργων, το ΕΦΣΙ και τα ομόλογα αυτά, τα οποία είναι δύο εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας ε, για να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη επενδύσεων. Ίσως ε, να σας ενδιαφέρει η ανακοίνωση που υιοθέτησε πολύ πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάνω στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Υιοθετήθηκε την 1η ε, Ιουνίου και στην ανακοίνωση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει ότι το φθινόπωρο θα υποβάλει περαιτέρω προτάσεις ε, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις στρατηγικές επενδύσεις όσον αφορά τα ομόλογα μεγάλων έργων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι θα πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα σε αυτά και τα ομόλογα δημοσίου χρέους, ε, τα οποία δεν είναι εργαλείο που βρίσκεται στη διάσταση της Ευρωπαϊκής διότι αυτό θα δημιουργήσει χρέος. Για να αποφύγουμε λοιπόν τις ε, παρεξηγήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι σύμφωνα με την ε, παρούσα συνθήκη οι διατάξεις ε, που έχουν να κάνουν με θέματα προϋπολογισμού και δημοσιονομικά έχουμε την αρχή της ισορροπίας που απαγορεύει τη δημιουργία ελλείμματος. Η αρχή αυτή επίσης ε, σημαίνει ότι πρόσθετοι πόροι δεν συνεπάγονται αναγκαστικά επιπλέον δαπάνες, διότι οι επιπλέον δαπάνες ε, θα πρέπει ε, να δημιουργούνται εντός του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Επίσης έχουμε την αρχή της οικουμενικότητας ε, που προβλέπει ότι τα έσοδα θα πρέπει να, να χρηματοδοτούν τις δαπάνες και δεν θα πρέπει συγκεκριμένα έσοδα να διατίθενται για συγκεκριμένες δαπάνες. Τέλος, ε, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει τη δυνατότητα να εισπράττει φόρους, ούτε να υποβάλει προτάσεις ε, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ευγνώμων για οποιαδήποτε συμβολή στην συζήτηση για το μέλλον της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πλαίσιο αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σεβαστεί πολύ αυστηρά την εντολή που συμφωνήθηκε στο τέλος των διαπραγματεύσεων για το προηγούμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, όπου τα τρία θεσμικά όργανα, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημιούργησαν ομάδα για ε, τους ίδιους πόρους, ε, τις οποίες προεδρεύει ο Μάριο Μόντι. Και περιμένουμε τις συστάσεις αυτής της ομάδας ε, μέχρι το τέλος του χρόνου και θα εξετάσουμε τότε εάν το σύστημα των ιδίων πόρων, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να τροποποιηθεί, διότι απαιτεί ομοφωνία όλων των κρατών μελών και επικύρωση σε όλα τα εθνικά κοινοβούλια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, θα εξετάσει όταν θα δημοσιευτούν οι ε, όταν λάβει τις συστάσεις της ομάδας Μόντι, ε, τι θα κάνει στη συνέχεια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Η κατάσταση είναι η εξή. Καταρχά είναι 6 και 4. Δεύτερον, ο αναφέροντας δυστυχώ δεν είναι παρόν. Τρίτον, είναι ένα περίπλοκο θέμα. Όμως, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι υπάρχει πρόβλημα και θα το παρακολουθήσει το θέμα αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να σας κάνω πρόταση, ειδικά προς τους σοσιαλιστές. Γιατί ήταν πρόταση των σοσιαλιστών να συζητηθεί το θέμα αυτό σήμερα. Κάνω λοιπόν την εξή πρόταση. Αν συμφωνούν οι συνάδελφοι, να κρατήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, θα περιμένουμε περισσότερε πληροφορίε από την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή δηλαδή Επιτροπή. Και τρίτον, να σταματήσουμε εδώ τη συνεδρίαση και να επανέλθουμε στο θέμα αυτό το φθινόπωρο. Συμφωνείτε? Γιατί μπορούμε να συνεχίσουμε την συζήτηση εδώ πέρα επαορίστο, μέχρι το... μπορούμε να μιλάμε αυτά μεσάνυχτα, χωρί τον αναφέροντα, χωρί να πετύχουμε τίποτα. Α περιμένουμε πληροφορίε, α κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά και το ξανασυζητάμε το φθινόπωρο. Συμφωνείτε. Well, I could talk on behalf of the petitioner. Να εκφράσω τη γνώμη του αναφέροντα. Γιατί ενεπλάκην στην σύνταξη της αναφοράς. Αλλά μια και η πρότασή σας είναι να αναβάλλετε την συζήτηση για το Σεπτέμβριο. Αυτό ήταν καταρχάς. Ναι. Ναι. Μέχρι το φθινόπωρο. Αν θα συμφωνήσουν βεβαίω και οι συντονιστέ με αυτή την επιφύλαξη. Γιατί μπορούμε να συνεχίσουμε να συζητάμε εδώ για ώρες. Αλλά θα είναι εντελώς αναποτελεσματική αυτή η συζήτηση. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και τεράστια χρονική πίεση εδώ. Παραμένει ανοιχτή αναφορά, περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κλείνουμε εδώ τη συνεδρίαση. Yeah, thank you, President. Um, of course... Ε, φυσικά. Δεν θα επιληθούν όλα τα προβλήματα σε σχέση με την αναφορά των πολιτών σήμερα. Ωστόσο το ζήτημα είναι πάρα πολύ επίκαιρο και σημαντικό και πιθανότατα θα εξεταστεί και σε άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή στο Κοινοβούλιο, την Επιτροπή Προϋπολογισμών, την εικόνα ακόμα οικονομική νομισματική, ακόμα και την Επιτροπή Πασχόλησης. <clears throat> Δεν είναι δυνατόν να σε σχέση με αυτή την αναφορά που κατέληξε σε αυτή την Επιτροπή να ακολουθηθεί άλλη διαδικασία. Θα πρέπει να εξεταστεί και από άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές και το φθινόπωρο να επανέλθουμε και να συζητήσουμε περισσότερο τα θέματα ουσίας. Συμφωνείτε, είναι καλή πρόταση αυτή. Βλέπω ότι υπάρχει μια τέτοια πρόταση και νομίζω οι συνάδελφοι συμφωνούν. Αυτό θα κάνουμε λοιπόν όπως αναφέρατε. Θα συμπεριλάβουμε και άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Ε, κυρία, εσείς θα ήταν δυνατόν να έχουμε την ευκαιρία συζητώντας ε, σε σχέση με τον, επίτροπο, με τον αναφέροντα να έχουμε αυτή τη συζήτηση ότι θα μπορούσαμε δηλαδή να είναι δυνατόν ώστε να εμβαθύνουμε σε αυτό το θέμα. Για να με Νομίζω ναι, θα μπορούσε να γίνει αυτό, ναι. Παρακαλώ εσύ συνάδελφε. Ε, Μια και μου δίνετε το λόγο, Πρόεδρε, να σου πω και εγώ δύο λόγια. Λέει ο κύριος Καλβέ Σομπού. Συμφωνώ με τον κύριο Γιώργο Λάινεν. Το γεγονός ότι θα εξεταστεί αυτή η αναφορά στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και Προϋπολογισμού ε, δεν θα πρέπει να καθυστερήσει η όλη διαδικασία, όπου και αν εξεταστεί. Μια και δώσαμε το λόγο όμω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νομίζω θα έπρεπε τουλάχιστον μέσα σε πέντε λεφτά να δώσετε το λόγο και στην εκπρόσωπο της ε, αναφέρουσα, να πει δύο λόγια, ούτω ώστε να απαντήσει και η Κομισιόν. Είναι πιο λογικό αυτό, πιο λογική διαδικασία. Υπάρχει συνένεση. Α, παραμένει ανοιχτή αναφορά. Θα ζητήσουμε περισσότερε πληροφορίε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα στείλουμε αυτή την αναφορά και στι άλλε αρμόδιε ε, κοινοβουλευτικέ επιτροπέ να μα πούν τη γνώμη του και θα ξανασυζητήσουμε με την παρουσία τη αναφέρουσα. Συμφωνείτε λοιπόν. Αυτή είναι η πρότασή μα. Παρακαλώ. Να διευκρινίσω κάτι. Γιατί ο κύριος Γιολάινεν αναφέρθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών Απασχόλησης και Προϋπολογισμών. Εγώ είμαι μέλος Επιτροπής ΕΜΠΛ, Απασχόλησης δηλαδή. Θα ήθελα οπωσδήποτε να στέλνει και στη δική μας Επιτροπή, να το τονίσω αυτό. Και θέλω να το επιβεβαιώσω. Πρότεινε ο κύριος Γιολάινεν, αλλά δεν ξέρω αν εσείς πρόεδρε συμφωνείτε να στέλνει και στη δική μου Επιτροπή. Ναι, ναι, το δεχόμαστε δεχόμαστε να σταλεί και στη δική σας Επιτροπή, στην Επιτροπή Απασχόληση. Επομένω, κλείνουμε εδώ, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ. Πρώτα ευχαριστώ και τους Γερμηνείς. Καλό σας βράδυ. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στι 9.